Επίσης, ε, η γνωμοδότηση τονίζει ότι η προενταξιακή βοήθεια θα πρέπει να χορηγείται με τέτοιο τρόπο την Κομισιόν, έτσι ώστε να προετοιμάζονται τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των δαπανών των διαφόρων ταμείων. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την οικονομική ικανότητα στο πλαίσιο τη πρόταξη και να ευθυγραμμίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες για την προενταξιακή βοήθεια σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Οικονομικής Ανάπτυξη. Η νομοδότηση αυτή ε, αφορά και το ε, πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας για την πολιτική γειτονία. Μία τροπολογία έχει κατατεθεί που ο είναι πρόθυμος να την δεχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. να άλλος, πώς έλεγε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης ηγητής, ε, συγκαστηρίζω την γνωμοδότηση του κ. Ρούτσεκ καθώς επίσης και την τροπολογία της συναδέλφου Ίνσκι που διευκρινίζει περαιτέρω τη γνωμοδότηση αλλά που πάει προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Οι καθυστερήσει όμως που συνεχίζουν να υφίστανται για την προταξική βοήθεια θα πρέπει να βελτιωθεί από την, ε, με, την δημιουργία ε, διοικητικών ικανοτήτων. Η Κροατία είναι μια χώρα που θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την επόμενη χρονιά. Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν με την έκθεση Ρούτσεκ και με την τροπολογία της συνάδελφου Νέμψκε. Θα ήθελα όμως να κάνω άλλη μια παρατήρηση που πάει πέρα από τη συγκεκριμένη νομοδότηση που μας απασχολεί. Να σας αναφέρω κάτι που με απασχολεί με ανησυχία. Είναι κάτι το οποίο θα έλεψε την προσοχή της Επιτροπής μας. Την περασμένη εβδομάδα ένα από τα δικαστήρια του Τσεχίας ε, κύρωσε την, την ένταξη της ε, ε, συγγνώμη, πρόκειται για τη Βουλή της Κροατίας που ενέκρινε την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, ε, εκτός από την Ιταλία, καμία άλλη μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κύρωσε την ε, ένταξη. Είχαμε πει ότι οι κυρώσεις θα έπρεπε να γίνουν πριν από την 31η Δεκεμβρίου. Τώρα όμως ε, ήδη ο Βρετανός πρόεδρος της Βουλής είπε ότι θα περιμένουν τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και θα ακυρώσουν την επόμενη χρονιά. Την 1η Ιουλίου όμως η Κροατία θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θεωρώ ότι είναι παράδεκτος διαδικασία. Εμείς ΑΦΕΤ, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα χρειαστεί να φροντίσουμε το συντομό των δυνατών κάποια από τα μεγάλη κράτη να κυρώσουν συμπεριλαμβανομένως και της χώρας μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που επανέρχομαι η δεύτερη φορά, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που αφορά στη χώρα μου. Υποχρεωμένο να πάρω τον λόγο λοιπόν. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η έκθεση Roadcheck είναι πολύ χρήσιμη. Ούτω ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι και κυρίως η Κροατία να επικεντρωθούν στα πιο σημαντικά θέματα, δηλαδή διαχείριση της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου με την ενταξιακή περίοδο. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί ε, το δυναμικό, το δυναμικό ε, και να παγιωθεί ε, ο τρόπος διαχείρισης της ενταξιακής βοήθειας. Όλα αυτά αναγνωρίζονται. Επίσης, όταν αποφασίσουμε τα ποσά που θα δοθούν ε, στην Κροατία στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας στην Κροατία, ε, ούτως ώστε να τη βοηθήσουμε να απτύξει αυτό το δυναμικό της. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν για την προετοιμασία την έκθεση, για τα συμπληρώματά τους και τις προτάσεις τους. η επιθυμία της Κροατίας είναι να είναι ένα καλό και αποτελεσματικό κράτος μέλος. Ευχαριστώ για την υποστήριξη σας, λέει ο κύριος Ζάλα. Ε, δεν έχω άλλα σχόλια. Μάλιστα. Νομίζω, όπως είπε ο κύριος Πόσελ, θα πρέπει να ακούσουμε κάποια πράγματα για τη διαδικασία επικύρωσης, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό θα ήταν, χρήσιμο θα ήταν να ενημερωθούμε σε ποια φάση είναι, να δούμε ποια είναι τα εμπόδια σε κάποιες χώρες που δημιουργούν μια διαδικασία ανάσχεσης. Θα σταματήσουμε τώρα για λίγα λεπτά. Γιατί περιμένουμε την κυρία Κοστολέβα και την κυρία Βίγκαν.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 the lady who made the report. Meine Damen und Herren, das ist zum Περνάμε τώρα στο σημείο 5 κυρίε και κύριοι τη ημερήσια διάταξη. Ο επικεφαλή αντιπροσωπή σε σχέση με τη Λευκορωσία, κ. Κάτσμαρεκ, δεν μπόρεσε να έρθει επίση λόγω του ποδοσφαίρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο. Όχι γιατί να λάβει καμιά προπόνηση, αλλά γιατί δυστυχώς πρέπει να πάει σε μια κηδεία. Πάντως, η κυρία Γιούλια Κοστελέβα είναι εδώ, την καλωσορίζουμε. Θα μας μιλήσει για τον αντίκτυπο των στοχοθετημένων κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως και βέβαια το έχουμε δει όχι μόνο όσον αφορά την Λευκορωσία, αλλά μας ενδιαφέρει και γενικότερα ως ζήτημα. Έχουμε πει στον κύριο Βίγκαντ εδώ, διευθύνοντα σύμβουλο τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Παρακαλώ λοιπόν, μια και έχουμε αρκετή, αρκετά θέματα να συζητήσουμε πιστεύω, την κυρία Κοροστέλεβα να λάβει το λόγο πρώτη για να μας κάνει την παρουσίασή της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρίε Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Έχω να σας παρουσιάσω σήμερα με την έκθεσή μου τη Γενική Επισκόπηση των ε, επιπτώσεων των στοχοθετημένων ε, κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή θα επικεντρωθώ σε κύρια θέματα που έχουν να κάνουν με κύριους οικονομικούς παράγοντες και τις συνέπειες αυτούς ε, στη Λευκορωσία, επιχειρήσεις κυρίως δηλαδή και αξιολόγηση των πιθανών κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας, δηλαδή πόσο με τα συμπεράσματα και συστάσεις. Η πολιτική καταστολή που ξεκίνησε το 1995 στη Λευκορωσία με την απόπειρα του Λουκασένκο να επεκτείνει τις, ε, να διευρύνει τις ε, προεδρικές του ε, εξουσίες και μετά το 1996 με το δημοψήφισμα με το οποίο προσπάθησε να εξασφαλίσει έγκριση του συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και με την υποκατάσταση του Κοινοβουλίου με μια κοινοβουλευτική συνέλευση που θα τον υπηρετούσε. Εν λοιπόν έχει ξεκινήσει μια πολιτική η οποία παγίως παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία και τις ε, πολιτικές ελευθερίες ε, μετά από τις προεδρικές εκλογές του 1900 του 2010, μετά 19 Δεκεμβρίου του 2010, που οδήγησε σε καταστολή εις βάρος της αντιπολίτευσης και σε καταπίεση και καταστολής βάρος των διαδηλωτών και απολύσεις εργαζομένων που είχαν ταχθεί κατά του καθεστώτος. καθώς και ε, μελών του Συμβουλίου από τη Εκπαίδευση Ευκορωσία. Εντέδασε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εισαγωγή κυρώσεων για την περίοδο μετά το 2010 απαγορεύσει ε, ταξιδε, ταξιδιών, εξαγωγών, πάγωμα οικονομικών στοιχείων, στοχευμένο καταρχά, σε συγκεκριμένα άτομα λόγω των, ε, των πολιτικών του πράξεων καταστολή στη Λευκορωσία Απαγόρευση ταξιδιού επίσης για ορισμένους επιχειρηματίες ε, προσκύμενους στο καθεστώς και τους φορείς που αυτοί έλεγχαν. Εκλήθην λοιπόν να εξετάσω καταρχάς αν ήταν αποτελεσματικές αυτές οι κυρώσεις για την ε, πολιτική αλλαγή στη χώρα, με στόχο την πολιτική αλλαγή στον χώρο και δεύτερον εάν θα είχε νόημα η διεύρυνσή τους ε, για να εξασφαλιστεί το ε, ευκταίο αποτέλεσμα. Η πολιτική των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Λευκορωσίας μπορεί, όπως έχει τώρα, να χαρακτηριστεί ως ε, πολιτική ευφυών κυρώσεων, στοχεύεται δηλαδή συγκεκριμένα άτομα, με προσπάθεια ταυτόχρονα και να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες για τον γενικότερο πληθυσμό Στο πλαίσιο λοιπόν των ευφυών κυρώσεων ε, γίνεται αυτό με στόχο, όπως είπα, να εντοπίζεται ποιος είναι υπεύθυνο υπέτειος για τις ε, μη αποδεκτές πολιτικές ε, και τακτικές στην Λευκορωσία και αντιστοίχως να επιβληθούν οι κυρώσεις περιορισμός, παραδείγματα στις προ... περιουσιακά του στοιχεία και ούτω καθεξής. μέσα σε δύο εβδομάδες περίπου από την εισαγωγή των ε, κυρώσεων και δι των ε, της απαγορεύσης ταξιδίου από την ε, Λευκορωσία κοίταξα ιδιαίτερως τα αγετικά στελέχη του καθεστώτος και τους οικονομικούς παράγοντες που πρόσφερε στο καθεστόν μέσα από μια δικτυακή πύλη ουκρανική η οποία από το 2007 παράγει μελέτες για την ε, επιχειρηματική ελίτ στην Λευκορωσία, καλύπτοντας πάνω από χίλια άτομα, χίλιους επιχειρηματίες. Ιδιαίτερος ωστόσο ε, ενδιαφέρον είχε η ταξινόμηση των πρώτων 200 σημαντικότερων ε, επιχειρηματιών της Λευκορωσίας. Για να εντοπιστεί λοιπόν αυτή η ελίτ, την οποία με δύο κριτήρια εντόπισα, την επιχειρηματική επιτυχία, κεφαλαιοποίηση στην αγορά δηλαδή, κυρίως των επιχειρήσεων και ε, επιρροή που μπορεί να ασκήσουν ε, μέσω της ε, διαπλοκής σε ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης. Επτά ήταν αυτοί οι οποίοι εντόπισα από την έρευνα αυτή. για τους οποίους ε, στοιχειοθετείται στενός δεσμός με τον ίδιο τον Λουκασέγκο και την οικογένειά του. Χωρίς λοιπόν να σας δώσω λεπτομερή στοιχεία για καθέναν από αυτούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαγάγει κυρώσεις κατά τριών εξ αυτών των επτά, το BTF, το CHISH και τον Τυρνάφσκι Ωστόσο, ο κατάλογος των ε, φορέων που έχουν περιληφθεί στον, ε, στη μαύρη λίστα τη λεγόμενη είναι πολύ ευρύτερος. Και αν θέλετε θα μπορούσα με τις ερωτήσεις σας να δώσω πιο πολλά στοιχεία για, τα, ε, για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επτά επιχειρηματίες. Όπως είπα τα κριτήρια ήταν η επιτυχία, η επιχειρηματική μεγαλύτερη συμβολή, το μεγαλύτερο ποσοστό της συμβολή στην ε, οικονομία της Λευκορωσίας και η διαπλοκή με την ε, ηγεσία της χώρας. Οι κύριες επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν ε, επίσης παρουσίαζαν σημαντικό δυναμικό σύμβασης, συμβολή στο ΑΕΠ και παραγωγή στι Και ήταν είτε η κατασκευαστική στις μηχανές, βέβαια απευθύνεται κυρίως στην Ουκρανική αγορά, το δεν έχει πολύ μεγάλη ε, δραστηριότητα στο εξωτερικό, η κατεργασία τροφίμων, επεξεργασία τροφίμων, πάλι για την ε, ρωσική αγορά και την ε, κοινοπραξία αναξιωτών κρατών, χημική και πέτροβιομηχανία με τον όμιλο Περνεύτυχημ που απευθύνεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ειδικότερα εξαγωγών ε, ορυκτών και χημικών. Και ως εκ τούτου παρουσιάζεται, εμφανίζεται ως η σημαντικότερη επιχείρηση, με βάση τα στοιχεία του 2011, με 39% έναντι του 34% που έχει η Ρωσία ε, στις εξαγωγές αυτές. Άρα έχουμε βασικά αγαθά, ορυκτά, ακατέργαστο και κατεργασμένο ε, πετρέλαιο. Βλέπετε ότι στη διαφάνεια μας έχουμε βάλει τα ποστά 36% για το 2011 και χημικά προϊόντα, κάλιο και λοιπάσματα. Όπως είπα, βασικά αγαθά λοιπόν που απευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συζήτηση λοιπόν σε σχέση με τις κυρώσεις περιορίζονται συνήθως στο κατά πόσο είναι αποτελεσματικές ή όχι κυρώσεις. Από πλευράς βέβαια της χώρας, <clears throat> από την οπτική γωνία της χώρας στην οποία επιβάλλονται, αλλά και σε σχετισμό με τη χώρα από την οποία επιβάλλονται. Κυρίως λοιπόν διαπιστώνεται ότι λιγότερο αποτελεσματικέ θα είναι σε περίπτωση ενός αυταρχικού καθεστώτος ή καθεστώτος οι γενικές κυρώσεις δεδομένου ότι μπορεί ε, η ηγετική ελίτ, η ηγετικη ΛΕΙΤ η ηγεσία να απαλλαγεί από τις δυσμένες συνέπειες αυτών και να τις μετακυλήσει στο γενικό πληθυσμό. Και έτσι θεωρήθηκε ότι θα πρέπει οι κυρώσεις να αφορούν είτε τις εξαγωγές ακατέργαστου του πετρελαίου, λιπασμάτων ε, κατεργασμένου πετρελαίου και οικονομικών ε, κινήσεων, κινήσεων κεφαλαίων Προ τη Λευκορωσία κυρίω, όχι προ τη Ρωσία δηλαδή και την κοινοπραξία, αλλά και θα, θα σήμαινε αυτό ότι θα μπορούσε η Λευκορωσία να αναζητήσει διαφορετικές οδούς, αλλά κινδυνεύει να χάσει το επενδυτικό της δίκτυο και μπορεί να αναγκαστεί να ιδιωτικοποιήσει στρατηγικούς φορείς και τόσο η Λευκορωσία όσο και η Ρωσία και ως εκ να αναζητήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα με τα δεδομένα αυτά θα μπορούσε να ωφεληθεί η γενικότερη η, ελίτ και το κόστος το κοινωνικό για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι πολύ πιο σοβαρό. Πράγμα το οποίο θα οδηγούσε ενδεχομένω και σε ενίσχυση ακόμη του καθεστώτος, δηλαδή θα έχει το αντίθετο από το επιδεκόμενο αποτέλεσμα. Και έτσι προτείναμε να εστιαστούμε περισσότερο, ως πιο βιώσιμη λύση, σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες υψηλό κόστος των συναλλαγών, δηλαδή για τις, ε, για τις ε, συναλλαγές τους, θα μειωνόταν η αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές και βέβαια αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αναδιανομή ωφελών ε, στους ανταγωνιστές τους που προκειμένου θα ήταν Ρώσοι επιχειρηματίες. Φυσικά αυτό λαμβανωμένο υπόψη είναι ότι δεν είναι οι μόνοι που συμβάλλουν στον ε, προϋπολογισμό της χώρας, αλλά πάλι μπορούν να στηρίξουν ε, με, τα, με τη χρηματοδότησή τους ε, την κυβέρνηση, το καθεστώς και το έχουμε δει αυτό πολύ συγκεκριμένα με την οικογένεια του Λουκασέγκο και τον Λουκασέγκο τον ίδιο, ο οποίος έχει πολύ στενούς δασμούς με ορισμένους από αυτούς τους επιφανείς, ούτως οι είναι επιχειρηματίες. Μια και δεν έχω χρόνο λοιπόν, αφήνω τα ε, αφήνω την ανάλυση και προχωρώ στα συμπεράσματα πιο συγκεκριμένα, όπως τα έχουμε καταγράψει, τις, στάσεις τις καλύτερα, για να πω ότι για λόγους συμβολισμού η απαγόρευση ταξιδιών θα πρέπει να συνεχιστούν, έχει, ε, ε, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτός, αυτή η απαγόρευση, ιδιαίτερα θα ήταν καλό εάν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή σε κατασταλτικές δράσεις ε, και άλλων προσωπικότητων, να επεκταθεί και σε αυτό. Το εμπάρκο σε όπλα μπορεί να έχει πάλι σημαντικό χαρακτήρα, αν και δεν, έχει, δεν φαίνεται να έχει διάθεση εμπόλεμη η Λευκορωσία. Η κυρώσεις που αφορούν κύριους επιχειρηματικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα γιατί είδαμε παραδείγματι πρόσφατα την αποφυλάκηση των υποψηφίων πρόεδρων των τελευταίων προεδρικών εκλογών του Σάνεκεφ και της Πατερένεκα και θα έλεγα ότι θα ήταν πρόημο μάλλον να ε, καταργηθούν κυρώσεις κατά των επιχειρηματιών όπως ο Πέφτιεφ, ο Τσίκ ε, και ο Τερνάυσκι. Υπάρχουν κάποιοι κρατούμενοι ακόμη, πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές που περιμένουμε να απελευθερωθούν. Άρα τέτοια ζητήματα και θέματα ακόμη αλλαγή του καθεστώτος δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. Επίσης, ένας, ε, μια μαύρη λίστα θα μπορούσε να περιλάβει τη προσωπικότητα που σα ανέφερα και νωρίτερα, να διευρυνθεί δηλαδή για να περιλάβει και άλλους. Και ω εκ τούτου χρειάζεται να ενισχυθεί η δέσμευση στράτευσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεργασία τη με το λαό της Λευκορωσίας και την κοινωνία των πολιτών, με υποστήριξη και οικονομική των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καλό δηλαδή να δοθεί εντύπωση ότι μόνο κατά της ηγεσίας ε, προστασίας της, ε, του καθεστώτος και κατά των πιο επιφανών επιχειρηματιών στρέφονται κυρώσεις αυτές και όχι κατά του γενικότερου πληθυσμού. Επίσης, ε, κλειδί της επιτυχίας για, για τις στοχευμένες αυτές κυρώσεις είναι η αποφασιστική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με τις κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει να στραφούν έστω και αν αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες ε, κατά των επιχειρηματιών. Ειδικότερα αναφέρομαι στη Σλοβενία και το Γιώζιτσις όπου ξέρουμε ότι είχε συμφέροντα οικονομικά επενδεδημένα η Σλοβενία και χρειάστηκε να διακόψει τους οικονομικούς δεσμούς με κάποιες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Περιμένω τις ερωτήσεις σας φυσικά και ευχαριστώ να δώσω απαντήσεις ό,τι σας απασχολεί πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Βίγκαντ και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συστήσω το θέμα των κυρώσεων εις βάρος της ε, Λευκορωσίας. Η συζήτηση φτάνει σε μια σημαντική χρονική στιγμή Έχουμε διάφορα ορόσημα μπροστά μας. Τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην ε, Λευκορωσία το Σεπτέμβριο και την ε, αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης των περιοριστικών μέτρων που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναθεώρηση που θα γίνει τον Οκτώβριο. Δυστυχώς ε, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ υπάρχει επιδείνωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών και φυσικά έχουμε εξακολουθούμε να έχουμε πολιτικούς κρατούμενους στη χώρα. Τους τρεις ε, πρώτους μήνες ε, του 2012 είχαμε ενίσχυση του καθεστώτος περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις να διευρύνει τα κριτήρια με βάση τα οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα, ούτως ώστε να τα προσαρμόσει στην αλλαγή του τρόπου εφαρμογής της καταστολής και να υπάρξει και μια ειδική νομική βάση, ούτως ώστε να εστιάσει κυρίως σε επιχειρήσεις που πρόσκειται στο καθεστώς. Ε, διευρύθηκαν τα νομικά κριτήρια λοιπόν για να καλύψουμε όχι μόνο την ε, καταστολή μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2010, αλλά και άτομα και φορεί που επωφελούνται ή που υποστηρίζουν το καθεστώς καθώς και άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ε, καταστολή της αντιπολίτευσης και της κοινωνία των πολιτών. Πέρα από τον ταξιδιωτικό περιορισμό που υπάρχει και, τον, και το εμπάργκο όπλων, μπορούμε να διευρύνουμε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που στοχεύουμε με το την ταξιδιωτική απαγόρευση, αλλά και για πρώτη φορά να έχουμε συγκεκριμένες ε, κυρώσεις κατά επιχειρηματιών. Αυτή είναι και η σύσταση που προκύπτει από την έκθεση της κυρίας Κοροστέλεβα. Στις 20 Μαρτίου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πήρε μια απόφαση πολύ συγκεκριμένη. Ήταν η πιο σκληρή απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο μέχρι στιγμής απέναντι στη Λευκορωσία και πιο σκληρή να προσθέσει στα περιοριστικά μέτρα και άλλα 12 άτομα. επιφανής ε, ε το της Ιντεράσκη και καθώς και 12 ε, επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς που προσθέσαμε στον κατάλογο αυτό. Ήταν δύσκολες αυτές οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών, γιατί βεβαίως αυτές οι κυρώσεις ε, έχουν και οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορα από τα κράτη-μέλη μας. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν διαφέρουμε σε τίποτα από τις κυρώσεις που επιβάλλουμε στη Συρία και στο Ιράν. Ε, Επίσης, οι αντιδράσεις από λευκορωσικής πλευράς ε, δείχνουν ότι πέρα από τον κύριο Πέφτη, ε, τα άτομα αυτά τα οποία συμπεριλάβαμε στο κατάλογο και οι επιχειρήσεις εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Επίσης, όπως τόνισε και η έκθεση του Κοινοβουλίου, ακούσαμε τη φιλοσοφία των, του Συμβουλίου που βασίζεται στην προσπάθεια να μειωθεί οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο γενικό πληθυσμό. Μια από τις βασικές επιπτώσεις τη έκθεσης αυτής του Κοινοβουλίου ήταν ακριβώς αυτή. Και επίση ένα παράδοξο που θέλω να το τονίσω είναι έχουμε επιβάλει αυτές τις κυρώσει μεν, αλλά παρόλα αυτά ε, αυξάνονται οι εξαγωγές αυξήθηκαν πέρυσι οι εξαγωγέ τη Λευκορωσία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 16,9%. Ενάμιση χρόνο μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Φεβρουαρίου πέρσι, 243 άτομα και 32 επιχειρήσεις έχουν μπει σε αυτόν τον κατάλογο, το πίνακα, το μαύρο κατάλογο τέλο πάντων. Ταυτόχρονα η κατάσταση στη Λευκορωσία το συγκεκριμένο αυτό χρονικό διάστημα επιδεινώθηκε περαιτέρω. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι τα περιοριστικά μέτρα ήταν αναποτελεσματικά, θα ήταν λαθασμένο συμπέρασμα. Αντίθετα, έχουμε την εκτίμηση ότι τα μέτρα μας που ήταν περιοριστικά ήταν πολύ σημαντικά πολιτικά για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Μίνσκ και εξακολουθούν να πιέζουν την κυβέρνηση γιατί η απόδειξη είναι η απελευθέρωση των 23 πολιτικών κρατουμένων που έγινε πέρυσι, 21 ε, απελευθερώθηκαν μεταξύ του Αυγούστου και του Οκτωβρίου 2011 και 2 τον Απρίλιο του 2012. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το Μάρτιο είπε ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι ανοιχτά ε, και είναι υποσυνεχή αναθεώρηση και το Συμβούλιο θα αναφέρει άτομα και επιχειρήσεις ε, και θα τα βάζει σε αυτόν τον κατάλογο όταν υποστηρίζουν ε, το καθεστώς, εκτός και αν απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να προσθέσω και δύο λόγια για την, κατάσταση, την ευρύτερη κατάσταση της Λευκορωσίας και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο ο Σανίκο και ο Μποναρέγκο ε, που ήταν πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν. Ήταν θετικά νέα αυτά, ευπρόσδεκτα και αμέσως μετά ε, στείλαμε πίσω του πρέσβεις μας ε, στο Μίνσκ. Αυτό δεν είχε σχέση με τις ε, απελευθερώσεις και ούτε είχε σχέση και με τις γενικές σχέσεις με την Λευκορωσία. Ήταν μια δράση η οποία έγινε με συντονισμό όλων των κρατών μελών. Αυτή η θετική εξέλιξη από την αρχή του Μαΐου ε, επέτρεψαν να μειώσουν κάπως τις εντάσεις μας στις διμερείς μας σχέσεις και να δημιουργήσουν ένα παράθυρο ευκαιρίας, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το ΜΙΣΚ. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση σε πολλούς τομείς είναι ανησυχητική. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, ακούμε ότι γίνονται παρενοχλήσεις ε, εκπροσώπων το, της κοινωνίας των πολιτών μέσω με κρατήσεις, με διοικητικές κυρώσεις κτλ. Ο, κύριο, ο κύριος Παρφιάνκοφ ε, απελευθερώθηκε γιατί κρατεί μετά τις ε, διαδηλώσεις ε, της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές. Αλλά ε, ξανασυλλήφθηκε γιατί υποτίθεται ότι παραβίωσε τους όρους της αναστολής του. Ο, ο νόμος για την Ε, δίνει περισσότερες ευκαιρίες, ε, στην, περισσότερες εξουσίες μάλλον στις ε, υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Πέρα από τους νόμους που επικυρώθηκαν πέρυσι για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την κοινωνία των πολιτών κτλ. Και ελπίζουμε οι αρχές Λευκορωσίας να μην πάρουν κι άλλα τέτοια μέτρα. Αυτό που θέλουμε είναι η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Ε, μας δίνουν κάποια μηνύματα ότι θα το κάνουν, αλλά δεν προβαίνουν ε, στην ίδια την πράξη. Θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ε, και να υπάρξουν ίσοι όροι α, στους οποίους συμμετέχουν όλοι στις εκλογές. Προς το παρόν, οι σχετικοί νόμοι της Λευκορωσίας δεν έχουν αλλάξει. Οι απελευθερώσεις ε, πολιτικών κρατουμένων δεν άλλαξαν το κλίμα στην, στο Μίσκ και ούτως ή άλλως το μπαλάκι παραμένει στο στρατόπεδο του Μίσκ. Ε, το θέμα δεν είναι να απελευθερωθούν κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι, όλοι πρέπει να απελευθερωθούν και θα πρέπει τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα να αποκατασταθούν πριν αλλάξει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση την πολιτική της και άρει τα περιοριστικά μέτρα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να έρθουμε σε επαφή με, τους, με την αντιπολίτευση, το κοινό, την κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία και με την έκθεση και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τονίσω δύο θέματα προς αυτό. Καταρχάς το θέμα της διευκόλυνση ε, των θεωρήσεων. Τον Ιούνιο του 2011 ε, προσφέραμε στην ε, Λευκορωσία να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την διευκόλυνση από το καθεστώ υποβολή θεωρήσεων. Αυτό αφορούσε γενικά τον πληθυσμό, είναι γενικά ένα ελκυστικό μέτρο για τι τρίτε χώρε, αλλά δεν πήραμε επίσημη απάντηση από το ΜΙΣΚ. Από επίσημε επαφέ, καταλαβαίνουμε ότι το ΜΙΣΚ δεν θέλει να διευκολύνει ε, τα ταξίδια για τον ίδιο ε, πληθυσμό τη. στο βαθμό που υπάρχουν 243 άτομα στον κατάλογο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λευκορώσοι, που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να αυξήσετε τις, ε, τα μονομερή μέτρα, τα κάτι μελη δηλαδή, στο επίπεδο αυτό. Επίσης, ε, ξεκινάμε ένα διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση για τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στην Λευκορωσία και για τις σχέσεις της Λευκορωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε στη Λευκορωσία για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μια προσπάθεια καινοτόμα, ε, το κάνουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και έχουμε τέσσερις ομάδες εργασίας που καλύπτουν ευρύ φάσμα δράσεων και μεταρρυθμίσεων. Έχουμε ε, εντυπωσιαστεί από την, ε, τις γνώσεις των συμμετεχόντων πλευράς Λευκορωσίας και έχουμε και θεματικά σεμινάρια. Το πρώτο έγινε στην Βαρσοβία για την, ε, τις ιδιωτικοποίησεις. Επίσης έχουμε τετραπλασιάσει τη βοήθειά μας προς την κοινωνία των πολιτών. Όλες αυτές είναι προσπάθειες για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο και να παρεμποδίσουμε την, τα περαιτέρω δυσμενή γεγονότα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Hvala lepa eh, za zanimivo eh, eh, in potrebno poročilo. Ευχαριστούμε για αυτήν την ε, παρουσίαση και τις προφορίες που μας δώσατε. Εκπροσωπώ την Σλοβενία και θα ήθελα να μάθω πώς, ε, τι συνέχεια δόθηκε σε αυτό το ζήτημα το οποίο εσείς δείξατε. εσείς. Κυρία Κοροστλέβα είπατε πως η Σλοβονία ε, εκπροσωπεί κάποια στρατηγικά συμφέροντα. Νομίζω πως ε, σε, αυτές σε αυτό το διαγωνισμό συμμετείχαν και άλλες χώρες πλην της Σλοβενίας. Εντάξει, η Σλοβενία κέρδισε το διαγωνισμό. Δεν θα αναφέρω ποιες άλλες χώρες συμμετείχαν, αλλά από ό,τι γνωρίζω στην ε, Σλοβενία δεν, ε, ε, δεν, δεν επηρεάστηκε από την, την κατάσταση και δεν υπήρχε κάποιο κάποια κύρωση το οποία έπρεπε να έτσι Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Από ότι παρακολούθησα στον τύπο για πρώτη φορά το ζήτημα των κυρώσεων συζητήθηκε κατά τη Γιουντίκ. Η, Σλοβενία ήταν αντίθετα. Ήταν αντίθετη σε αυτή την απόφαση. Εξετάστηκε ένα επενδυτικό σχέδιο. Η Λευκορωσία Στη Λευκορωσία πρόκειται για το ξενοδοχείο Καμπίνσκι, το οποίο θα συμμετείχε, στην κατασκευή του οποίου θα συμμετείχαν ε, Σλοβαίνοι. Και ε, πρόκειται να λάβουν την υπεργολοβία. Κοιτάξτε, η όλη διαδικασία των κυρώσεων κατά κάποιων επιχειρηματιών ήταν κάτι το οποίο είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Γιούντιτσιτς που είναι ένας ε, επιχειρηματίας ε, συμπεριλήφθη στον πίνακα των επιχειρηματίων τους οποίους στόχευαν οι κυρώσεις ε, οι η Σλοβενική κυβέρνηση το εξέτασε και ζήτησε να υπάρξουν αποδείξεις σχετικά με την ε, συμμετοχή του Ιουδιτσιτς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα εξετάζεται ή μάλλον επανεξετάζεται. Το ίδιο αφορά, ε, το ίδιο αφορά και στον Αντώλη Τσορνιέσκη. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Συνεχίζω, κύριε κύριος Μπέλντερ, συγγνώμη που έφτασα με κάποια καθυστέρηση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Το κείμενο του Βίκτορ Μάθιουβιτς το διάβασα και αφορά την άποψη των, του συγγραφέα σχετικά με την συμπεριφορά των υπηρεσιών ασφαλείας και τη δράση τους κατά των αντιφρονούντων ή κατά ατόμων τα οποία εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα και διερωτώμεθα τι επιρροή μπορούμε να ασκήσουμε για να ζητήσουμε από τις αρχές της Λευκορωσίας να μην αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο τους πολίτες. Ε, ακόμα και όταν έχουν αντίθετες ε, θέσεις, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, π.χ. το διαδίκτυο, το οποίο εδώ και μερικά χρόνια χρησιμοποιείται για να καταγγείλουν κάποια πρόσωπα. Οι πολίτες διαβάζουν σχόλια τα οποία τους αφορούν και τα οποία έχουν συντάξει αυτές οι υπηρεσίες. Εξάλλου προσωπικότητες οι οποίες θεωρούνται από τις αρχές της Λευκορωσίας ως ανικαθεστατικοί, ε, κινηματογραφούνται και δημοσιεύονται αυτές οι εικόνες ε, ακόμα και να αφορούν την προσωπική τους ζωή και τον ιδιωτικό τους βία. Και πραγματικά διαρωτώ με τι πίεση μπορούμε να ασκήσουμε προς τα όργανα ασφαλείας, ε, ΚΑΓΕΜΠΕ, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες ασφάλειας του Λουκασέγκου. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Έρχεται, είναι στον δρόμο από το αεροδρόμιο. Ούτε αυτός τα κατάφερε. Ο κύριος Μπέλερ ήταν θαραλέος, γιατί από το όλμησε να υπερασπιστεί και την Ολλανδία στο ποδόσφαιρο. Έχετε τίποτα κύριε Βίγκαντ εσείς? Η κυρία Κωστόλεβα. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι το μήνυμα που είπε σήμερα ο κύριος Μπέλτα γεννά πολλές ανησυχίες. Οι συνάδελφοι στο Μίνσκ βλέπουν με θλίψη τους πόσο πιο αποτελεσματική γίνεται μέρα με τη γέρα, μέρα η μηχανή της καταστολής. έχουν τελεπορθεί και οι ξένοι διπλωμάτε. Βέβαια, καμία σύγκριση με τα όσα περνούν οι άνθρωποι που επιδεικνύουν το θάρρο το οποίο επιδείξατε εσεί, το οποίο μάλλον περιγράψατε εσεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να γίνουν σημαντικέ μεταρρυθμίσει τόσο στο πολιτικό όσο και το οικονομικό επίπεδο. Και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον ότι αυτή η κοινωνία αλλά και πολλοί εκπρόσωποι της ε, αντιπολίτευση θέλουν να αναλάβουν μαζί με την Ευρώπη τα απαραίτητα εκείνα βήματα που θα τους επιτρέψουν να ξεπεράσουν την, ε, το αδιέξοδο, την ακινησία σε σχέση με ε, τα προβλήματα αυτά πολιτικά αλλά και οικονομικά, δηλαδή να προχωρήσουν προς την ιδιωτικοποίηση στη χώρα τους ώστε να ξεκινήσουν και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα λένε ότι θα πρέπει και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως να εμπλακούν στη συζήτηση στο βαθμό που είναι δυνατόν, ώστε να υπάρχουν, ε, μάλλον ε, εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού θα πρέπει να υπάρχουν στην ε, προσπάθεια αυτή, στο διάλογο, ώστε να υπάρχουν και εκείνοι που γνωρίζουν την ουσία των πραγμάτων σε πυρογνώμονες, εκπρόσωποι λοιπόν του κρατικού μηχανισμού, οι οποίοι θα μπορούν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όπως αυτά στα οποία αναφερθήκατε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε στην ε, προσπάθεια αυτή και στον ε, δρόμο αυτόν και τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης. Α, όχι, παρακαλώ, εσείς ε, θέλατε κάτι να συμπληρώσετε, κυρία Κορόστλεβα. Πάντως θέλω να πω ότι με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθήσαμε την εκθεσή σας, την παρουσίαση και η μέθοδος και οι πληροφορίες που μας δώσετε ήταν πάρα πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Ξέρουμε, όσο παραδεκτό και αν είναι, ότι συνεχίζεται η ποιήση βάρος διαφορών οργανώσεων και φορέων στην Ουκρανία και των και ενημέρωσης. Οργανωμένη πίεση και αφόρητη πολλές φορές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το και να μας παρασύρει σε λάθος αποτελέσματα. Σας ανθαρρύνω να συνεχίσετε το έργο σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προχωρούμε στην κατάσταση στην Ουκρανία και τις προοπτικές της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Όχι το ίδιο ακριβώς, αλλά πάντως είναι κατεύθυνση το θέμα. Και θα ακούσουμε τις απόψεις των παριστομένων, αλλά πρώτα ο κύριος Τάνοκ θα κάνει την εισήγηση. Μετά ο κύριος Α, όλοι οι Πολωνοί φίλοι απουσιάζουν σήμερα. Ο κύριος Κόβαλ, ο κύριος Κούτκο. Θα πρέπει να είναι κλεισμετό το αεροδρόμιο στη Βαρσοβία φαίνεται. Αστείο, αστείο ήταν αστείο. Mr Mr. Uh, uh, colleague, uh, Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λεκούτκο Κάπου έχει πιαστεί σε μποτιλιάρισμα από ό,τι φαίνεται. Είναι στον δρόμο πάντως, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, αλλά είναι στον δρόμο. Και μου ζήτησε το μεταξύ να διατυπώσω για τον κύριο Βίγκαντ εκ μέρους του κάποιες ε, ερωτήσεις. Και μια και τις ε, έλαβα μόλι πριν από λίγο. Ελπίζω να μπορούσα να τι εκφράσω σωστά. Λοιπόν, κύριε Βίγκαν, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι ακριβώ η εξέλιξη προ την διαδικασία τη ε, Συμφωνία Συνδέσεω και τι ακόμα στάδια μένουν μέχρι την τελική υπογραφή. Επίση, τι, διαθέσει εκδηλώνει το Συμβούλιο έναντι τη ε, Συμφωνία Συνδέσεω και τη ε, κατάσταση προκύπτει από την φυλάκιση τη Γιούλια Τιμοσέγκα. Τι προϋποθέσεις αναμένουν ε, τα κράτη-μέλη να εκπληρώσει η Ουκρανία πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως και τι εναλλακτικέ επιλογές υπάρχουν. Εάν αυτές δεν πληρωθούν, επίσης ε, μπορεί να αναβληθεί επαόριστον αυτή η Συμφωνία Συνδέσεως ε, και να παραμείνει ενισχύει η τρέχουσα Συμφωνία Εταιρικής Οικονομικής Σχέσης και επίσης τι μπορεί το Κοινοβούλιο ή τι θα κάνει το Κοινοβούλιο μέχρι ότου λάβουμε τελικά το κείμενο της συμφωνίας, τι σχέδια υπάρχουν ως προς την υλοποίηση της συμφωνίας συντάσεως με, συντάσεως με την υπογραφή της από τα κράτη-μέλη, τι τμήματα της συστάσεώς μας υλοποιήθηκαν ή έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω ή τι σκοπεύει να υλοποιήσει από αυτά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω στου προσοχής μείνουν αυτά εκ μέρους του καθηγητού Λεκούτικο ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει εγκαίρως για τις συνεδρίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Παρακαλώ, κύριε Βίγκαντ. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Τάνακ, για τις πολυόρθμες αυτέ ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν μπορώ επαρκώς να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Προφανώς και οι εξελίξεις ε, στην Ουκρανία στους προσεχείς μήνες και οι αποφάσεις που θα ληφθούν ε, ε, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Μετά από την τελευταία συνάντηση στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Ποπόσκι, ε, Γενικού Γραμματέα και ο, και ο κ. Φιούλε συναντήθηκαν με τους ευρωβουλευτές Νομίζω ότι είναι και η ώρα να ξανασυζητήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την Ουκρανία. Ε, καλωσορίζουμε την μελέτη για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανία. Σημειώνουμε τις πολλές επισκέψεις που έκαναν οι Ευρωβουλευτές τις τελευταίες εβδομάδε στην Ουκρανία ε, και ε, την πρωτοβουλία του Προέδρου Σούλτ μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Αζάροφ, τον Πρωθυπουργό, το Μάιο, Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης για τον διορισμό του κ. Πέτκοξ ε, και την, τον παρατηρητή που αποστήλαμε από πλευράς Πολωνικής Πολωνίας μάλλον, για να παραστεί στη δίκη της κυρίας Τιμοσέγκο. Η εντολή των, δύο προέδρων μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει και περιπτώσεις ε, του κυρίου ε, Εύαρη Βασένκο και του κυρίου Λουτσένκο. ούτως ώστε όλες οι περιπτώσεις ε, επιλεκτικής δικαιοσύνης να παρακολουθηθούν. Πριν αντιδράσω στις ερωτήσεις σας, κύριε Τάνοκ, Θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να ακούσετε και κάποια σχόλια που αφορούν την κατάσταση της Ουκρανίας και τις προοπτικές που έχει στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης. Στα μέσα του Μαΐου, πριν από το Συμβούλιο Συνεργασίας, ε, κάναμε μια συζήτηση προσανατολισμού μεταξύ των 27 Υπουργών Εξωτερικών για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία, δεδομένης πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε και το νέο ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία στις 24 του Μαΐου. Επίσης, η Ουκρανία σταδιακά μπαίνει στην περίοδο προεκλογικής εκστρατείας. Θα γίνουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές ε, τον Οκτώβριο και θα είναι η Λιβύα για μας για να αποτιμήσουμε το βαθμό με τον οποίο οι, βαθιές, αρχές σέβονται τις δεσμεύσεις τους ότι οι εκλογές θα γίνουν με βάση τα διεθνή πρότυπα. Έχουν προσκαλέσει τους περισσότερους νατούς παρατηρητές από την ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ε, οι οποίοι θα εξετάσουν ε, το κατά πόσον είναι δίκαιες και ανώθευτες οι εκλογές αυτές. Ε, όχι μόνο κατά τη μέρα των ε, διεξαγωγής των εκλογών, αλλά και την προεκλογική περίοδο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με την Ουκρανία και υπάρχει πλήρη συνεννόηση μεταξύ των θεσμικών εργάτων της εργοάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 30 Μαρτίου ε, μονογράφηκε η Συμφωνία σύνδεσης και έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει την οικονομική ένταξη της Ουκρανίας και την πολιτική της ένταξη και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να υπάρξουν νέες οικονομικές ευκαιρίες σημαντικές, αλλά και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία. Μπορεί να μετασχηματίσει λοιπόν και την κοινωνία και την οικονομία αν εφαρμοστεί σωστά. Ε, μονογράφτηκε η συμφωνία από τους βασικούς διαπραγματευτές και είναι το πιο φιλόδοξο κείμενο που έχει προετοιμάσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το απευθύνει προς μια τρίτη χώρα. Με βάση ε, τις κοινέ αξίες που μοιράζονται και οι δύο πλευρές και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Θα προσεγγίσει η Ουκρανία ε, το κοινοτικό κεκτημένο, το ενωσιακό κεκτημένο και θα εξυγχρονιστούν οι θεσμοί της και θα ανέβουν τα πρότυπα διακυβέρνηση της χώρας. Τι περιμένουμε από την Ουκρανία ούτω ώστε να δουλέψει αυτή η συμφωνία. Είναι η πρώτη και συγκεκριμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προβληματικές επιπτώσεις της επιλεκτικής δικαιοσύνης, όπως ε, συνέβη στην περίπτωση της Τούλιας Τιμοσέγκο και άλλων. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Επίσης, θέλουμε να διεξαχθούν οι βουλευτικές, ε, κοινοβουλευτικές εκλογές με βάση τα διεθνή πρότυπα. Δεύτερον και τρίτον, να προχωρήσουν πολλές καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις που είχαμε συμφωνήσει 7 χρόνια πριν με την Ουκρανία και που συνοψίζονται στην συνοψισμένη ε, ατζέντα ε, σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η Συμφωνία Σύνδεσης που συμπεριλαμβάνει και την ζώνη ελευθέρου εμπορίου ε, βαθιού και ευρέως εμπορίου. Σε αυτή τη συμφωνία σύνδεσης εμείς παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εσωτερικές εξελίξεις στην όμορη χώρα ιδίω τις διάφορες δίκες εναντίον μελών της πρώην κυβέρνησης, την περίπτωση Τιμοσέγκο βέβαια, αλλά και του πρώην Υπουργού Εσωτερικού Λουτσέγκο, του πρώτη ε, υπουργού, ε, πρώην Υπουργού Άμυνα Τιμωσέγκο ε, και περιβάλλοντος Φιλιτσούκ. Όλοι αυτοί είναι σήμερα φυλακισμένοι, σε κράτηση. Θέλουμε ε, να προχωρήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά μας στην, ε, στη σχέση με την Ουκρανία και πιστεύουμε ότι είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ να κρατήσουμε μια εστιασμένη προσπάθεια διαλόγου με το Κίεβο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς και κάποια συγκεκριμένα θέματα όπου πιστεύουμε ότι τώρα τα καταφέρνουμε. Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο. Ε, μας... Υπάρχει μια στρατηγική για την ε, μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημοσίων ε, οικονομικών που προωθεί η Ουκρανία και αν γίνει κάτι τέτοιο θα ξαναρχίσει η χορήγηση ε, βοήθειας για τη στήριξη του προϋπολογισμού. Επίσης, η δέσμευση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Υπάρχει σχετικός διάλογος. Επίσης, η Ουκρανία είναι ανοιχτή για να ξαναρχίσουν ε, συζητήσεις για τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου και να προχωρήσουν οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις για την αυτογκάζ. Επίσης, ε, θα πρέπει να εκμοντερνιστεί ο τρόπος διαμετακόμισης του φυσικού, ε, φυσικού αερίου. Υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου προχωράει η προσπάθεια, όπως στα πλαίσια της, της, του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων, ε, και με αυτόν τον τρόπο κρατιέται ζωντανή η σχέση μας με την Ουκρανία. Η εκπαίδευση, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, ε, το περιβάλλον, εκεί δεν υπάρχει πρόοδος όμως. Φυσικά μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο σε πολλούς τομείς, αλλά τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν, τα ανέφερα, είναι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και η υπόθεση των δικών και της επιλεκτικής δικαιοσύνης. Όποια και είναι τα αποτελέσματα στις εκλογές και στις μεταρρυθμίσεις, πιστεύουμε να προχωρήσει η Ουκρανία, να μην μας δώσει απλώς εξηγήσει, να κάνει βήματα. Οι δίκες ε, των πολιτικών της πρώην κυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν με δίκαιο τρόπο. Μέχρι στιγμής ε, δεν είχαν γίνει με βάση τα διεθνή πρότυπα, οι δικαστές δεν ήταν αδέκαστοι, ε, δεν, ήταν, δεν είχαν τα ίδια όπλα η εισαγγελία και η υπεράσπιση. Το θέμα δεν είναι οι προσωπικότητες, οι πού πρόσκειται ο καθένα, αλλά το θέμα είναι ε, εγγενές, είναι διαρθωτικό. Ε, ο κώδικας ποινική δικο... θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί, δεν έχει μεταρρυθμιστεί, σε στενή συνεργασία ε, με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει να, είναι να ήταν σε κράτηση ε, μέχρι τη δίκη τους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σωστή παροχή ιατρικής βοήθειας για την Τζούλια Τιμοσένκο. Αλλά και αυτή δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Επίσης υπάρχει ένας νέος κώδικας ποινική δικονομίας, ε, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να υπάρξουν δίκαιοι δίκη, δίκες δίκες στο μέλλον. Περιμένουμε να υπάρξει συμπληρωματική νομοθεσία για να εφαρμοστεί αυτός ο νέος κώδικας, δηλαδή νόμοι για το πώς διεξάγει το έργο του ο εισαγγελέα, ε, οι δικαστές, ε, να μεταρρυθμιστεί το καθεστώς των δικαστών και όλες αυτές είναι συστάσεις που έχουν γίνει από την Επιτροπή της Βενετίας. Όποιο και είναι το πολιτικό κλίμα στην Ουκρανία, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, χρειάζονται ε, παραταξιακή στήριξη, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα συστημικά προβλήματα, τα διαφορετικά προβλήματα που έχουμε δει στη λειτουργία του συστήματος της δικαιοσύνης αποκατασταθούν και ότι οι πολίτες εποφελούνται ε, από όλε αυτές τις δικαστικέ μεταρρυθμίσει, αν εφόσον εφαρμοστούν πλήρω. Πριν περάσω τις ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις της Συμφωνίας Σύνδεσης, θα ήθελα να πω ότι τα όσα διέρευσαν από το γραφείο της εισαγγελία ε, δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ε, όπως είπε και ο Επίτροπος Φιούλε την περασμένη εβδομάδα, το να δικάζεται κανείς από τα ΜΜΕ ε, είναι παραβίαση της δικαιοσύνης. θα, θα παρατηρήσουμε τις, ε, την εξαγωγή των υπόλοιπων δικών με καλή προσοχή. Επίσης, θέλουμε να ολοκληρωθεί το των δυνατών τεχνική δουλειά για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Ε, χαιρόμαστε που μονογράφτηκε η Συμφωνία και η τεχνική και νομική αναθεώρηση του ενωπημένου κειμένου ε, έχει προχωρήσει. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς, και μιλάμε για 1.200 σελίδες περίπου, έτσι, είναι ότι τώρα έχουμε επιτάπητος ένα από τα πιο φιλόδοξα κείμενα και τις πιο περίπλοκες συμφωνίες που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα. Φυσικά θέλουμε αυτή η προσπάθεια να μην πάει χαμένη. Θέλουμε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία που μονογράφηκε. Η υπογραφή της συμφωνίας θα απελευθερώσει ένα δυναμικό για πλήρη εξυγχρονισμό και μεταρρύθμιση της χώρας και θα δημιουργήσει συνένεση στη χώρα. Θα ήταν καλό για την Ουκρανία, θα ήταν καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θα είναι καλό για την, συμφωνία, την Ανατολική Συμφωνία Τελικής Σχέσης. Η απόφαση για την υπογραφή όμως της συμφωνίας έγκυται στα χέρια του Συμβουλίου και θα γίνει επί τη βάση των κριτηρίων τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Ε, κοινοβουλευτικές εκλογές, ε, επιλεκτικές δίκες και μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας με την Κομισιόν θα, θα υποβάλει ένα σχέδιο πρότασης για υπογραφή όταν τεχνική δουλειά ολοκληρωθεί και επί τη βάση της αξιολόγησης των προϋποθέσεων το Συμβούλιο θα λάβει την τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσει και θα περάσει στην υπογραφή της συμφωνίας ή όχι. Φαντάζεστε ότι η διάθεση στο Συμβούλιο, όπως είπατε και εσείς, αφορά για το χρόνο της υπογραφής της συμφωνίας. Ε, η διάθεση δεν είναι αυτή, δεν κινείται προς, την, προς μια κατεύθυνση, δεν είναι συνενετική απόλυτα, γιατί εξαρτάται φυσικά από τις ε, εξελίξεις στην Ουκρανία. Αν οι τρεις προϋποθέσεις που ανέφερα πριν ε, υπάρξουν, και αν υπάρχει ένα θετικό κλίμα για να προτείνουμε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής της σύνδεσης, τότε θα το προτείνουμε η Ουκρανία να γνωρίζει ότι η συμφωνία ούτω ή άλλως δεν θα υπογραφεί πριν από τις εκλογές και δεν γίνεται να υπογραφεί πριν από τις εκλογές. Η Επιτροπή Άφετη υποστηρίζει και υποστηρίζει πάντα το κράτος δικαίου, την δημοκρατία στην Ουκρανία, καθώς και τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον μαζί σα προ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά το μπαλάκι είναι στο Κίεβο για να δούμε πόσο γρήγορα και πόσο μακριά θα πάμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Βίγκαντ. Λίγο χρόνο έχουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν μαζί τις ε, τρεις παρεμβάσεις για να απαντήσετε μετά μου. Ο εισηγητής Country Monitor. Παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς, κύριε τον Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βίγκαν που ήρθε ανάμεσά μας και μας μίλησε για αυτά τα ζητήματα που όλο και περισσότερο διεθνοποιούνται Όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας ε, είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι διότι γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό είναι ζωτική σημασία για την ε, Ουκρανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προχωρήσει η Συμφωνία Σύνδεσης και η Ουκρανία να συμμετέχει σε αυτήν την ευρία συμμαχία των δημοκρατικών κρατών. Αυτές οι ελπίδες όμως, αυτές οι προσδοκίες δυστυχώς του τελευταίους μήνες παρεμποδίστηκαν ε, από τα τεκτενόμενα και δεν ξέρουμε τι μπορούμε να προσδοκούμε στο, για το εγγύς μέλλον. Το κείμενο αποτελείται από 1200 σελίδες και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν κάποια τμήματα που μας δείχνουν ε, μια κάποια πρόοδο, αλλά γενικά οι μεταρρυθμίσεις, ε, οι εκλογές, ε, και η επιλεκτική δικαιοσύνη είναι τα θεμελιώδη του κράτους δικαίου και πιστεύω ότι όλη αυτή η πρόοδος ε, που επιτέθηκε μέχρι τώρα αφορά σε μια πρόοδο η οποία όμως ε, δεν ε, μας κάνει να ελπίζουμε σε κάτι το ιδιαίτερο θετικό τους προσεχείς μήνες. Εσείς ε, πολύ προσεκτικά αποφύγατε να απαντήσετε στο θέμα του χρονοδιαγράμματος αλλά θα ήθελα κάποιες πληροφορίες περί αυτού και με την ενδεχόμενη δυνατότητα άσκησης ε, μόχλευσης ως Ευρωκοινοβούλιο για να επιταχύνουμε τα πράγματα διότι δεν είναι προς το συμφέρον μας η κατάσταση στην Ουκρανία να επιδεινωθεί περαιτέρω και ελπίζω πως κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ μπορώ να πω ότι συμμορώ, συμπερίζομαι συνολικά τις ε, αξιολογήσεις. Πρέπει νομίζω τώρα να ομολογήσουμε ότι και το θέμα της δικαιοσύνης και η διεξαγωγή των ε, εκλογών ε, θα είναι το αντιδραστήριο από το οποίο θα κριθεί η πορεία αυτής της ε, κυβέρνησης. Το κείμενο μεταρρυθμίσει όσο ωραία λόγια και να έχει και όσο ωραία σχέδια και να περιλαμβάνει, εάν δεν υλοποιηθεί δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήθελα να επισημάνω σε κάποιες επαφές που είχα ε, άκουσα από τους Ουκρανούς ότι όχι μόνο στο Λινμπέρκ αλλά και στο Χάρκιφ μπορεί να υπάρχουν υποψήφοι της αντιπολίτευσης η οποία, η οποία ούτως είπε προληπτικός ε, φυλακίστηκαν, κατηγορήθηκαν για κάποια άσχετα δικήματα και προληπτικώς μπήκαν στη φυλακή προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στις ε, προσεχείς εκλογέ. Ε, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει. Πρέπει να το εξετάσουμε με σοβαρότητα. Για τους κύριους Κρασινεύσκη και το Κόξ Ίσως η συνέντευξη αυτή του κυρίου Κρασνιέσκη στην Γκαζέτα Βιμπόσκα δεν ήταν πολύ καλή ιδέα τη προηγούμενη εβδομάδα η συνέντευξη. Δεν έχει κανένα λόγο να κάνει σχόλια για το ποιο μπορεί να, να ε, κερδίσει τι εκλογέ. Και σε τελευταία ανάλυση και εκείνο ω τελευταίο κομμουνιστή υπουργό, καλό θα ήταν με το ιστορικό αυτό τέλο πάντων να αποφεύγει σχόλια. Βλέπουμε ορισμένου όπως αυτός ε, που έχουν πολύ στενούς δεσμούς με ε, ολιγάρχες, ε, οικονομικά συμφέροντα ε, να έρχονται μετά εδώ και να σχολιάζουν, να επικρίνουν διάφορα κόμματα χωρίς όμως να είναι ήδη πραγματικά υπέρμαχοι της δημοκρατίας. Κύριο Κρασνεύσκη, καλό θα ήταν να ήταν πολύ πιο μετρημένος και να απέφευγε τις δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερω για την ε, παρουσία με την οποία παρουσιάσατε κύριε Σούλτ, την, ε, ε, τον αγώνα για, την, το κάτω δικαίου στην Ουκρανία με την κυρία Χάρμς. Έχετε το λόγο. Ναι, πρόεδρο, δεν έχω ερωτήματα. Είναι πολύ σωστή, ήθελα να πω, πολύ εύστοχη η παρουσίαση του κυρίου Βίγκαντ. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι μας ε, επέτρεψε να επισκεφθούμε την κυρία Τιμοσένκο, να μιλήσουμε μαζί της, ε, να μιλήσουμε και με τον Υπουργό και θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες της κυρίας Τιμοσένκο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Τιμοσένκο, χαίρετε ιδιαίτερος για την αλληλεγγύη που επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σαφή τοποθέτηση, ε, κυρίως από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συγκεκριμένα, ε, παρακολουθεί λοιπόν τι εξελίξει κυρία από την, από την ε, τηλεόραση, έστω και από το κρεβάτι στο νοσοκομείο, στο οποίο βρίσκεται. παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και από ό,τι φαίνεται και από τις ε, δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτη στις επιλογές των ψηφοφορών, παρότι έχει ξεκινήσει και μάλιστα διεξάγεται κατά τρόπο όχι καθαρό η προεκλογική εκστρατεία, γιατί γίνονται προσπάθειες και δωροδοκίας και πίεσης προς τους υποψηφίους. Γι' αυτό θα ήταν καλό το ταχύτερο δυνατό να α, παρέμβουμε, να προσπαθήσουμε να πείσουμε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ε, μάχη επικράτησης, γιατί εάν ε, ξεκινούσε μία διαδικασία ψήφου δυσπιστίας φαρους του ε, Προέδρου θα κινδύνευε να χάσει και την θέση του. Άρα γίνονται πάρα πολλέ προσπαθίε χειραγώγηση του αποτελεσματικού των εκλογών. Η κυρία Τιμοσέγκο έχει επιδείξει πολύ μεγάλο θάρρος ε, η, η, απέστειλε επιστολή και στην κυρία Μέρκελ ευχαριστώντα γιατί και οι ιατροί της ε, φιλανθρωπικής οργάνωσης Αριτέ, η κυρία Χάρμς ε, και άλλοι ήρθαν ε, σε επαφή μαζί της, της προσέφεραν και γιατροφαρμακευτική περίθαλψη ε, και έτσι βρίσκεται μέσα σε ένα νοσοκομείο, σε μια μάλλον νοσοκομιακή ιατρική μονάδα φυλακών υπό καθεστώς πολύ αυστηρής παρακολούθησης. Έχει κάμερες μέσα στο ίδιο το δωμάτιο στο οποίο είναι κλινήρης, υφίσταται ψυχολογικό πόλεμο και τρομοκρατία. Προφανώ μέσα σε συνθήκε οι οποίε δεν συμβαίνουν καθόλου στη βελτίωση ε, των συνθήκων ε, τη υγεία τη. Και βλέπουμε ότι όπως και ο Πούτιν είχε κατηγορήσει τον Ροτοκόφσκι για απόπειρες, ε, απόπειρα φόρνου και δεν είχε κανέναν τρόπο να απαντήσει στην, ε, στις κατηγορίες. Έτσι και η κυρία Τιμωσέγκο βρίσκεται κατηγορούμενη για ε, διάφορα και ποικίλα εγκλήματα. Για δε την γενικότερη πολιτική θα ήθελα να πω ότι οι Συμφωνία συνδέσεις βέβαια τη πάρα πολύ η Ουκρανία, αλλά χωρίς ελευθερία και δημοκρατίες. Δεν νομίζω ότι έχει για μας τουλάχιστον νόημα μια τέτοια συμφωνία σύνδεσης. Και πες περιπτώσει καλό θα ήταν ίσως ε, να δούμε πώς μπορούμε να όπως το χωρίσουμε, να είπα να χωρίσουμε καλύτερα χωρίς όμως να ε, χαθούν και τα προσχήματα. Το πιο σημαντικό σε σχέση με την κυρία Τιμοσέγκο είναι ότι η ίδια υπογραμμίζει ότι έχει λιγότερη σημασία η δική της η μοίρα, η δική της η τύχη από ότι άλλους, άλλων ε, πολυάριθμων, ε, ανώνυμων και πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχουν διάφορα φαινόμενα ευνίδιας ε, ασθένειας όπως μιας παράξενης μορφής υπατήτηδας η οποία έχει προσβάλει ε, Κάποιου ε, κρατουμένου, χωρί ακριβώς να ξέρουμε, αλλά με πολύ σοβαρέ επιπτώσει στην υγεία, χωρίς ακριβώ όμω να ξέρουμε πώ εμφανίζει. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχουν υπόνοιε για δηλητηρίαση και ούτω καθεξή. Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσουν τις προσεχεί μας προσπάθειες. Η κυρία Κορνέλισεν. Thank you. Um, thank you very much. Ευχαριστώ για τις προφορίες ε, που μας δώσατε για την επιλεκτική δικαιοσύνη. Διαρωτώ με και για κάποια άλλα πράγματα που αφορούν στην Ουκρανία. Στις 20 Μαΐου έκανα ό,τι μπορούσα για να συμμετάσχω στην η παρέλαση στο Κίεβο ακυρώθηκε, αλλά έμαθα ότι κάποιοι συμμετέχοντες ε, <clears throat> κυνηγήθηκαν και οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν ε, να προστατεύσουν τα μέλη. Τώρα στο Κοινοβούλιο συζητείται ένας νόμος ε, κατά των ε, ομοφιλοφίλων και εάν περάσει αυτή η νομοθεσία τότε θα προβλέπουν ε, πολύ βαριές κυρώσεις Νομίζω ότι εδώ παραβιάζονται κάποιες ε, βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ελευθερία της έκφρασης, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη ως συντονίστρια της ομάδας ALDE να πω πως ε, συμφωνούμε με την ε, άποψη που εξέφρασε ο Βίλαντ και καθώς επίσης και με όλη την προσέγγιση. προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται επιλεκτική δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερα λεπτό. Γνωρίζετε αναβίβολα πως ο Γκίφερ Χόφστατ, ο πρόεδρος της Άλντε και όπως και ο κύριος Χάνς Πανμπάλε, πρόεδρος της Διεθνούς των Φιλελευθέρων, μετέβηκαν στο Κίεβο και είχαν συζήτηση με την Τζούλια Τίμοσενκο και ανέφεραν, ε, μας μετέφεραν μάλλον τις δύσκολες ε, και σκληρές συνθήκες ε, σύμφωνα με τις οποίες κρατείται στο νοσοκομείο. Χάνεται λοιπόν της απόλυτης στήριξής μας ως πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ. Well, thank you very much for your... Ευχαριστώ για την υποστήριξη σας, για την προσέγγιση μας Βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τις αξίες της πολιτικής γειτονία και της πολιτικής ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ε, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε με τους εταίρους που έχουν υψηλές φιλοδοξίες και που θέλουν να αποκτήσουν ε, βαθύτερη σχέση μαζί μας. Η ησυχία, η ησυχία λέει τι μόχλευση ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, χώρα αυτή. Την έχουμε και την ασκείτε κι εσείς, κρατώντας ένα πολύ αυστηρό έλεγχο. Εμπλέκεστε και πάρα πολύ από εσά προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια. Αν τελικά φτάσουμε όπως ελπίζω να φτάσουμε στη φάση προσωρινής εφαρμογής ε, από το Συμβούλιο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπογραφεί αυτή η εφαρμογή, άρα θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Ο Επίτροπος Εμπορίου είπε ότι παρότι δεν προβλέπεται στη συνθήκη, παρόλα αυτά θα έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν κάνει μια τέτοια πρόταση στο Συμβούλιο για να προχωρήσει ή όχι. Σε ό,τι αφορά την επικύρωση επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που έχετε. Η επικύρωση θα είναι μια διαδικασία με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι Ουκρανοί γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει θέση σε ισχύ, χωρίς να αλλάξει η πολιτική κατάσταση, χωρίς να πείσουν τα δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ε, χώρες μέλη, ότι έχει βελτιωθεί η πολιτική και η νομική κατάσταση στην Ουκρανία. Και για να απαντήσω πολύ στο στον κύριο Προφανώς με ένα νέο, μια νέα πυρική δικονομία δεν θα είχαμε 100% επιτυχία, αλλά πάντω χωρί νέα ποινική δικονομία δεν θα είχαμε καθόλου επιτυχία. Η οικονομία, ξέρετε, τη Ουκρανία είναι από την εποχή τη Σοβιετική, όπω και σε άλλα πρώην μέλη τη Σοβιετική Ένωση. Επομένω, έχουμε να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο, πρόοδο την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό, την οποία δεν, έχουμε δεν είχαμε εξασφαλίσει από την προηγούμενη κυβέρνηση και έτσι λοιπόν ε, ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας και με άλλα νομοθετήματα αλλά όπως είπατε πολύ σωστά πολύ σημαντικό είναι και το θέμα του διορισμού των δικαστών, των εισαγγελέων, υλοποίηση δηλαδή εφαρμογή αυτών των νέων ε, δικονομικών κανόνων και πάνω απ' όλα αυτό θα κριθεί στις ε, πολύ ενδιαφέρουσες για την, ευρία, για την ευρύτερη κοινή γνώμη αυτές δίκες. Επίσης, τα δικαιώματα της μειοψηφία. Πρέπει να πούμε ότι παραβιάζονται. Ανησυχητικές είναι οι συνθήκες στο Κίεβο. Η κοινότητα των ομοφιλοφίλων και, μετα... και φιλομεταβατικών παρεμποδίζονται δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ε, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα όταν παραβιάζει τα δικαιώματα. Είπα ότι εκπρόσωπο ε, έκανε δήλωση για αυτό το θέμα και εκφράζοντα την ανησυχία τη. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλου ότι για τι διακρίσει, στα πλαίσια του σχεδίου δράση για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων, υπάρχει προπόθεση για ευρία νομοθεσία που θα πρέπει να υπάρχει στην τρίτη χώρα και η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που υπάρχουν ε, στις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην ε, νοσιακή νομοθεσία κατά της, ε, των διακρίσεων γενικά. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και το θάρρος για να περάσει αυτή η νομοθεσία και πρόσφατα στη Μολδαβία είδαμε πόσα χρήματα έπρεπε να ξοδευτούν τόσο ώστε να περάσει ένας νόμος για την ισότητα χαιρετίζουμε την κυβέρνηση που πέρασε αυτό το νομοσχέδιο παρά την σημαντική αντίσταση από πολλές πολιτικές δυνάμεις. Ελπίζουμε αυτό να γίνει και σε πολλές άλλες χώρες, ανατολικές, ανατολικούς γειτόνους μας, ε, όπου συμφωνήσαμε μαζί ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοια βήματα ε, στα πλαίσια του καθεστώτος απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Φίγκαντ και αγαπητοί συνάδελφοι για τη συζήτηση, επιτρέψτε να κάνω παρατηρήσει. Ευχαριστώ τον πρόεδρο κύριο Κόξ για την ε, προσοχή και σύνεση που επιδεικνύει κατά την εκτέλεση των καθηκόνων του. Η διαδικασία βέβαια αυτή αφορά ολόκληρη την ε, έντολη. Δεύτερον, ε, συμφωνώ με τον κύριο Βίγκαντ όπως και πολλοί άλλοι. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε ενδιαφέρον το ταχύτερο δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία, να υπογραφεί και να τεθεί σε εφαρμογή. Και όπως είπατε, κύριε Βίγκαντ, είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο με διάφορα ψηφίσματα και συστάσεις του έχει ταχθεί υπέρ της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Τώρα το θέμα είναι ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ουκρανού Προέδρου. Θα δούμε αν ξέρει να παίζει μπάλα. Και όπως επεσήμανε και ο κ. Σούλτς νωρίτερα, η επιλεκτική αυτή δικαιοσύνη πολλές φορές έχει περιφερειακή υλοποίηση. Δεν αφορούν δηλαδή τα προβλήματα μόνο την κυρία Τιμοσέγκο, αλλά και πολλούς άλλους επιφανείς πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Ε, δηλαδή ποια είμαστε αντιμέτωποι και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι υποψήφοι της αντιπολίτευσης ε, στην επαρχία η πίεση που τους ασκείται προκαταβολικά, προληπτικά, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε εκλογές. Είναι πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι εκλογές ε, δεν χαρακτηρίζονται ως ε, ε καθαρές εκλογές ε, εάν την ημέρα των εκλογών πάνε όλα καλά. Καθαρές είναι οι εκλογές ε, ανώθευτες είναι εκλογές εάν μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι υποψήφοι και να συμμετάσχουν στην προεκλογική εκστρατεία συνολικά. Δεν μετράει δηλαδή μόνο η μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, δεν, μετράει μόνο η μέρα στην οποία ο πολίτης πάει στην κάλπη. Πρέπει να παρακολουθήσουμε ολόκληρη αυτή την περίοδο. Και πάντως, όπως είπα, για μια καλή εξέλιξη θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει ώστε να μην πάρει η Ουκρανία λάθος δρόμο. Λάθος δρόμο ο οποίος θα έφερνε ε, ε, και λάθος επιλογές ως προς τα δικαιώματα των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίγκαντ. Σας εύχομαι. Κάθε επιτυχία. Βλέπω πάντως ότι ήρθετε στο ύψος των περιστάσεων και των καθηκόντων σας.